ενεργό συμμετοχή τους και για τη βοήθησή τους και ελπίζω ότι όλοι αναμένουμε να παραβρεθούμε στη Βαλέτα όταν θα κοπεί η κορδέλα και θα εγγενιαστεί η υπηρεσία. Εγώ. Κλείνει η συζήτηση. Και δεν πρέπει να, να ξεχάσουμε ότι για 14 χρόνια προείδρευσε ε, αυτή τη συνεδρίαση ο συνάδελφός μας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές κυβερνήσεις το Βέλγιο, η Αυστρία συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 40 χρόνια. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου στη Μήνη Ολομέλεια. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης που είναι η έκθεση Κυριλόφ για τις γενικές διατάξεις του ΕΤΠΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Ταμείου Συνοχής για την ε, απλούστευση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση. Ο εισηγητής, ο κύριος Κυρίλοφ, είναι από αυτούς που μπλοκαρίστηκαν και δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο Στρασβούργο εξαιτίας ε, της ε, έκρηθμης κατάστασης της εναέριες μεταφορές. Και γι' αυτό η κυρία Κρέλ θα λάβει το λόγο εξ του κυρίου Κυρίλοφ. Κυρία Κρέλ, έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. λυπάμαι που δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα εδώ ο κύριος ε, κυρίλοφ γιατί εργάστηκε σκληρά για το θέμα. πρόκειται για θέμα που αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες και τις περιφέρειες της ένωσης. θα σας διαβάσω τώρα τις σημειώσεις του που είναι γραμμένες στα αγγλικά παρόλο που είναι βούλγαρος. Και επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις αλλαγές για τα ταμεία. Αυτές οι τροποποιήσεις προκύπτουν μεταξύ από τις κοινέ προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Είναι συνέχεια των εγγράφων που εγκρίναμε πέρυσι. Τότε είχαν γίνει... Κωνσταντς, οι διερμηνείς ζητούν να επιβραδύνεις λίγο για να μπορούν να σε παρακολουθήσουν. Με συγχωρείτε, δεν το κατάλαβα. Ζητώ από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να εργαστούν για την απλοποίηση των κανόνων για τα διορθωτικά ταμεία και για την αλλαγή των κανόνων έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις όταν το χρειάζονται τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω ότι υιοθετήθηκαν οι προτάσεις για απλοποίηση. Πιστεύω ότι οι αλλαγές που απλοποιούν κάποιες διατάξεις πρέπει να τύχουν της υποστήριξής μας. Μειώνεται το περιττό διοικητικό άγχος δημιουργείται μεγαλύτερη διαφάνεια και επιτρέπεται ο καλύτερος έλεγχος και οι λιγότερες ε, παρατυπίες. Αυτό σημαίνει καλύτερη δαπάνη των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για παράδειγμα, μέσω της τροποποίησης του άρθρου 87 ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να διορθώνουν τις παρατυπίες πριν βρεθούν από τα όργανα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κράτη-μέλη δεν χάνουν αυτά τα κονδύλια και θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για άλλα προγράμματα εντός του συνολικού προγράμματος. Μια δεύτερη τροποποίηση αφορά τις προκαταβολές για τις χώρες όπου είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κρίση θα υπάρξει αύξηση για το 2010. Επίσης όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλλού κονδύλια τα οποία δεν είχαν προλάβει να εγκριθούν ή να υλοποιηθούν εντός των προθεσμιών. Εξαιτία της σημασίας ενδεχομένως. Και επίσης υπάρχουν και μέτρα κατά της κρίσης που αυξάνουν την αλληλεγγύη και θα επιτρέψουν την ε, δαπάνη τη δημιουργία φρέσκων κονδυλίων που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά για την αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης των υποδομών και για την προσαρμογή των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε όλους τους τύπους μέτρων και θα είναι όλο και πιο χρήσιμα αν τα εφαρμόσουμε εγκαίρως. Δυστυχώς υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στο Συμβούλιο προκειμένου προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία όταν ήταν υπεύθυνο για την έγκριση του διορθωτικού κανονισμού. Πιστεύω ότι τώρα που το Κοινοβούλιο έχει εξίσου την αρμοδιότητα μαζί με το Συμβούλιο δεν θα αναβάλουμε περισσότερο την εφαρμογή αυτών των σημαντικών μέτρων. Θα μιλήσω τώρα εκ μέρους ε, του εαυτού μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους ε, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και Απασχόλησης που ασχολήθηκαν από το θέμα. Ελπίζω να μπορέσουμε να το εγκρίνουμε το Μάιο. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο τον κύριο Χάμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κυρία Κρέλ, σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση και επίσης σας ζητώ να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μου και στον κύριο Κυριλόφ γιατί γνωρίζω ότι όντως ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του σε αυτή την έκθεση. Μας επέτρεψε να περάσουμε γρήγορα από όλα τα θεσμικά εμπόδια και έτσι μπορέσαμε τώρα να έχουμε σε έναν κανονισμό που ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπερψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υλοποιηθεί άμεσα. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό παράδειγμα επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου και επίσης ένα καλό παράδειγμα του πώς η διάδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων μπορεί να έχει απτά αποτελέσματα. Γνωρίζω ότι θα έχουμε μία μακροπρόθεσμη απλοποίηση των κανόνων εξαιτίας αυτού του κανονισμού, ο οποίος ελπίζω ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί άμεσα και να ανακουφίσει έτσι τα κράτη-μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Για το λόγο αυτό είμαστε ευγνώμονες στο Συμβούλιο για την συμβιβαστική πρόταση που από ό,τι βλέπουμε τη στηρίζει μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού. Ουσιαστικά ένα θέμα του κανονισμού είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων και η απλοποίηση των σχετικών κανόνων. Πρόσφατα Δημοσιεύθηκε η πρώτη στρατηγική έκθεση για τα προγράμματα. Τώρα, λοιπόν, γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Δεν ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα για το τελευταίο εξάμεινο του προηγούμενου έτους, αλλά βελτιώνονται τα πράγματα και βεβαίως υπήρχε και το πρόβλημα των πολλών κανονισμών που έπρεπε να εφαρμόζονται παράλληλα. Ελπίζω λοιπόν ότι ο παρόν κανονισμός θα βοηθήσει την απλοποίηση αλλά και την μείωση του αντικτύπου της οικονομικής κρίσης. Ουσιαστικά, μέσω αυτού του κανονισμού Καταρχάς θα έχουμε ένα κοινό όριο 50 εκατομμυρίων για όλα τα προγράμματα. Επίσης θα είναι πιο απλή η διαδικασία για τις αιτήσει για προγράμματα, κάτι που θα απλοποιεί την όλη διαδικασία. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και την αντιμετώπιση της κρίσης καθώς και θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά για τη θέρμανση κτηρίων. Πέντε χώρες, Ρουμανία, Ουγγαρία και οι χώρες της Βαλτικής αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Ο νέος κανονισμός θα τους επιτρέψει να απορροφήσουν πιο γρήγορα κονδύλια και να τα δαπανίσουν πιο γρήγορα μέσω μιας πιο ευέλικτης εφαρμογής άμεσα θα υπάρχουν διαθέσιμα 750 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή προχρηματοδότησης και αυτό θα επιτρέψει σε πολλά προγράμματα να υλοποιηθούν γρηγορότερα. Επίσης, να πω ότι το 2009 6,2 δις δόθηκαν σε προχρηματοδοτήσεις και αυτό μας δείχνει ότι οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων μπορούν να δαπανηθούν άμεσα και όχι να δίνονται την τελευταία στιγμή. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή ομαλή χρήση τους και κάτι τέτοιο θα μπορέσει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Τώρα, θα παρεύουν οι ομιλητέ εξ ονόματο της Επιτροπής ε, αλλά ο κύριος Γκοτμάνη δεν τον βλέπω τουλάχιστον. Δεν είναι παρόν. Η κυρία Μπάστος λοιπόν έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Και εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα ήθελα να χαιρετήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο παρόλο που λείπει διότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την κυρία Κρέλη για την παρουσίαση που μας έκανε. Ο βασικός ε, στόχος είναι να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και να επιταχύνουμε ε, την δράση του ΕΤΠΑ και των κοινωνικών ταμείων. Άρα, στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής ε, κρίσης υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, η οποία θα μειωθεί όταν υπάρχει καλύτερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν φτάσουν αυτά αυτές οι επιδοτήσεις αυτούς που τις χρειάζονται. 20 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι, 4 εκατομμύρια περισσότεροι από ό,τι πέρσι και βεβαίως με ανωδική τάση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτό το βασικό μοχλό βοήθειας στην πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα της ΜΜΕ και την απασχόληση. Η ΜΜΕ είναι ο μοχλός της οικονομίας, η ατμομηχανή της ε, βιομηχανίας και της κοινωνίας. Χρειάζεται λοιπόν συνεχής απλούστευση και διασάφιση των νόμων που διέπουν την πολιτική συνοχής, κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο στη συζήτηση των προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με την συνεργασία των περιφερειακών κρατικών και τοπικών αρχών για να ορίσουμε καλύτερους κανόνες και λιγότερο γραφειοκρατικός για να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην ε, ε, εφαρμογή των προγραμμάτων μας. Ευχαριστούμε την κυρία Πάστος. Τώρα το λόγο έχουν οι ομιλητές που παρεμβαίνουν εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, των έξι ομάδων. Οι πέντε είναι κυρίες. Την κυρία Κονή δεν τη βλέπω. Ε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από μήνε και μήνε εργασιών, συλλογικών εργασιών, με πολύ επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή κύριο Κυριλόφ, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω δημόσια από εδώ. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να τονίσω την ποιότητα της εργασίας που επετέλεσε μαζί με το Συμβούλιο υπό την Ισπανική Προεδρία. Αυτό είναι σημαντικό διότι σήμερα συζητούμε για κανονισμό του οποίου τα μέτρα τα αναμένουν χιλιάδες άνθρωποι. Είμαι πεπισμένη ότι η περιφερειακή πολιτική είναι η διάσταση της Ένωσης που μεταφράζεται καλύτερα στην καθημερινή πράξη των ανθρώπων, των πολιτών. Έχει όμως την τάση να θεωρείται από όλους ως πολύπλοκη και αφηρημένη. Αυτή η εικόνα θα αλλάξει με την απλοποίηση των κανόνων που ζητούμε. Τα 350 δισεκατομμύρια των ταμείων υπάρχουν για να εξυπηρετούν τον πολίτη. Και αναμένουμε από τη μεταρρύθμιση να αποφέρει πραγματικά αποτελέσματα, ιδίως στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, παραδείγματος χάρη για να περιοριστώ σε ορισμένα μόνο θέματα. Περισσότερη ευελιξία και περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Περισσότερη ευελιξία διότι τα μέτρα απλοποίησης που προτείνονται επιτρέπουν τη μείωση των απαιτουμένων πληροφοριών και δικαιολογητικών και άρα μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερο κόστος, αλλά και μεγαλύτερη αλληλεγγύη διότι προβλέπονται έκτακτα μέτρα κατά πολέμηση των επιπτώσεων της κρίσης το είπε και η Επιτροπή και ένα νέο σύστημα υπολογισμών. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει τον Μάιο και έτσι θα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τα διαστροτικά ταμεία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι χρειάζονται ακόμη πάρα πολλά να γίνουν ως απλοποίηση. Ευχαριστούμε εξ των σοσιαλιστών. Το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Κάντενμπαχ. Κάλενμπαχ, με συγχωρείτε. Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη ότι ο Επίτροπος συνόψε πολύ καλά το όλο θέμα. Πρόκειται για ταχεία βοήθεια για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, αυτή την τρίτη αναδιατύπωση για τα διαρθρωτικά ταμεία, για να ανταποκριθούμε στην ε, δημοσιονομική κρίση, στην χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι τα διαρθρωτικά ταμεία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της περιφέρειας. Αυτό μας το δείχνει η πείρα μας. Και αυτό αφορά και τις ε, μελλοντικές προοπτικές. Θα πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιου τύπου κρίση, γιατί εμείς είμαστε οι πυροσβέστες της κρίσης. Περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για ευελιξία και αλληλεγγύη. Θα πρέπει να καταπραίνουμε, να μετριάσουμε την κρίση. Γι' αυτό χρειάζεται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτές τις προπληρωμές έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Αυτό το τόνισε και ο εισηγητής διαστόματος της κυρίας Γκρέλ. Άρα η μελλοντική πολιτική συνοχής θα πρέπει να σκιαγραφηθεί κατά τον, με τον κατάλληλο τρόπο για την ταχεία εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι δέχομαι ε, να τεθεί σε εφαρμογή τάχιστα αυτός ο κανονισμός. Εξονόδος των φιλελευθέρων. Η κυρία Μανέσκου έχει το λόγο, η οποία λάμπει δια της απουσίας της. Άρα περνάμε στους πρασίνους. Η κυρία Σρέτερ έχει το λόγο για τρία μισή λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, ας είμαστε απόλυτα σαφείς. Η απλούστευση την οποία όλοι για την οποία όλοι τα υπέρ όταν μιλάμε για αποχετευτικά, για αποτεφρωτήρες. Δεν ξέρω ε, κατά πόσο μπορεί να γίνει ένας τέτοιος παραλυσμός, αλλά πώς μπορούν να ε, προωθηθούν 25 εκατομμύρια, διότι μιλάμε για ένα κατόφλι 50 εκατομμυρίων. Αυτό που λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι η Κομισιόν δεν πρέπει να κάνει μια ανάλυση κόστους ωφελίας. Δεν θα διενεργηθεί καν μία τέτοια ανάλυση για ε, προγράμματα κάτω των 50 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Και κανένας, ε, κανένας έλεγχος δεν θα γίνει για να δούμε κατά πόσο ευθυγραμμίζονται αυτά τα προγράμματα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Άρα δεν θα γίνει κανένας τέτοιος έλεγχος. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να υπάρχει τέτοιο άχθος δανεισμού για τις περιφέρειες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα δαπανηθούν αυτά τα δάνεια για τις ε, τράπεζες. Ε, αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, διότι κατά τα πρώτα χρόνια θα ορίσουν πολύ ψηλά ε, επιτόκια για να χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται μελέτες ανάλυσης κόστους ωφελίας και πιστεύουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενδυναμωθεί και όχι να αποδυναμωθεί αυτή η τάση. Είμαστε κατά του κατοφλίου το οποίο ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια πλέον. Η ανάλυση κόστους ωφελίας θα πρέπει να γίνεται ανοιχτά και δημόσια για να ξέρουμε ότι συμβαδίζουμε και με τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Επίσης, ο κανονισμός λέει ότι ορισμένα προγράμματα ισχύουν, έχουν πενταετή διάρκεια. Εμείς οι πράσινοι μιλάμε για μία δεκαετή περίοδο, επέκταση δηλαδή σε δέκα χρόνια, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η επένδυση και να χρησιμοποιηθούν και να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Γιατί αν έχουμε πενταετή προγράμματα μόνο, δεν επαρκούν. Είχαμε την ε, περίπτωση της Νόκια στην ε, Βόρεια Βεσφαλία και βλέπουμε πώς έχει αυτή η προσέγγιση τη στιγμή που γίνεται ένας επιμερισμός αυτών των επενδύσεων. Θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα, να ορίσουμε μία ε, ρήτρα βιωσιμότητας 5 συν 5 και όχι μόνο τρία χρόνια όπως ναι. αναφέρει ο κανονισμός. Εμείς οι πράσινοι όταν μιλάμε για γενόδες επενδύσεις χωρίς ανάλυση κόσοφελίας θεωρούμε ότι αυτό ε, ενθαρρύνει την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος που πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Εάν δεν περάσουν οι τροπολογίες μας τότε δεν θα υπερψηφίσουμε τον κανονισμό. Επίσης ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία έτσι ώστε να δούμε αργότερα ποιος ε, ψήφισε υπέρ του κανονισμού. Γιατί ήδη δεχόμαστε παράπονα από τους πολίτες ότι προβαίνουμε σε κατασπατάληση χρημάτων και θέλουμε να ξέρουμε ποιος το προωθεί αυτό. Ο κύριος ε, Βανίστερο μας έδειξε την μπλε του κάρτα. Δεν ξέρω τι εννοείται ακριβώς γιατί μερικοί δεν γνωρίζουν τον κανονισμό και δείχνουν την ε, μπλε κάρτα για να εγγραφούν στο Catch the Eye. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βανίστερόι, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον κανονισμό, θέλει να υποβάλει μία ερώτηση στην κυρία ε, Σρέτερ. Κυρία Σρέτερ, δεχόσα την ερώτηση του κυρίου Βανίστερόι. Κύριε Βανίστερόι, έχετε το λόγο για να υποβάλλετε την ερώτησή σας. Θα ήθελα να πω ότι η συνάδελφος έχει αρνητική προσέγγιση στην ανάλυση της. Η αποκέντρωση των αρχών δεν είναι θετική μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής. Αυτό ακριβώς δεν επιθυμείτε, την αποκέντρωση αυτή έτσι ώστε μέσω συγχρηματοδότησης να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Γιατί σκιαγραφείτε τόσο αρνητικά την κατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος. Κυρία Στρέτερ, θέλετε να απαντήσετε πολύ σύντομα. Ναι, θα ήθελα και εγώ να απαντήσω. Αναφέρομαι σε μεγάλα σχέδια και προγράμματα μέσα στα πλαίσια μεγάλων επενδύσεων. Μιλάμε για 50 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία έχουν ελεγχθεί. Θα πρέπει όμως να δούμε που ε, διαθέτουμε τα χρήματα του φορολογούμενου. Διότι πολλές φορές γίνονται υπέρογγες επενδύσεις και ο φορολογούμενος καταβάλει το τίμημα. Ο κύριος Βλάσακ έχει το λόγο. Εξ ονόματος των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Είναι παρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε εδώ ένα συμβιβαστικό κανονισμό για αυλοποίηση της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρόκειται για κοινό στόχο και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2014. Οι προτάσεις αφορούν τα μεγάλα έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών σε θέματα ενεργειακής ε, αποδοτικότητας και αύξησης της ε, και μείωση μάλλον της ε, κατανάλωση ενέργειας για την θέρμανση κτίριων. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τροποποιήσουμε το υπάρχον σύστημα. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πρόκειται για συμβιβασμό και εδώ θα ήθελα να πω ότι στηρίζω την δήλωση της Ουγγαρίας που ζήτησε να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο τον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Δεν συμφωνώ με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την αποδέσμευση πληρωμών. Θεωρώ ότι οι ε, ε, ενισχύσεις θα έπρεπε να εγκριθούν εντός του 2010 Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν πολλές διευκρινήσεις. Παρόλα αυτά, εφόσον καταλήξαμε σε συμβιβασμό, πρέπει να κλείσουμε εδώ τη συζήτηση. Για εμένα το σημείο κλειδί είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία για τα διαρθρωτικά ταμεία και για τα κονδύλια που εγκρίνονται εδώ στο Στρασβούργο. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εργαστούμε σκληρά στις περιφέρειές μας. Εδώ θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες που έγιναν στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, στην Τσεχία που απλοποίησε ιδιαίτερα τις διαδικασίες για την ε, χρήση των κονδυλίων θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, διαχείριση και τον έλεγχο και τον έλεγχο παρατυπιών. Τώρα θα ήθελα να πω ότι η κυρία Ένς έχει το λόγο για τρία λεπτά εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, γιατί μιλάτε εξ ονόματος των ομάδων, μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ και εγώ εκπροσωπώ άλλους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν σήμερα. Καταρχάς, όσον αφορά την απλοποίηση της χρήσης των διαρθρωτικών κονδυλίων. Συμφωνούμε με αυτό το θέμα. Βεβαίω υπάρχουν κάποιες επικρίσεις όπως ανέφερε και η κυρία Σρέντερ. Παρ' όλα αυτά εμείς επικροτούμε την απλοποίηση και θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτός ο κανονισμός. Γιατί χάσαμε πολύ χρόνο σε συζητήσεις. ο συμβιβασμός που έχουμε μπροστά μας δεν ήταν αυτός που αναμέναμε αρχικά και έχουν αλλάξει πολλά από την αρχική πρόταση της προ... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το 100% για τις ε, προκαταβολές. Αυτό το μέτρο τελικά δεν συμπεριελήφθη και είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας να πω ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2009 είχε συζητηθεί κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το ερώτημα είναι, κάναμε αρκετά. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα διορθωτικά κονδύλια για καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης και για βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών των κονδυλίων. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτά τα κονδύλια είναι όντως σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και πρέπει να θυμόμαστε επίσης τις μεγάλες συνέπειες που είχε η κρίση στην αγορά απασχόλησης στην Ευρώπη. Έχουν αυξηθεί πολύ οι άνεργοι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανεργία και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με μεγάλους αριθμούς ανέργων. Και όλα αυτά θα είναι ανεξάρτητα από την κρίση. Οπότε η πρόταση της Επιτροπής αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα βήμα προς το εμπρός. Γιατί θα υπάρξουν και πέντε κράτη-μέλη που θα λάβουν σημαντική στήριξη. Πρόκειται για κράτη-μέλη στα οποία το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 10% ή περισσότερο μετά το 2008 και τα οποία πλέον θα μπορέσουν να λάβουν ιδιαίτερη στήριξη από το Ταμείο Συνοχής. Επαναλαμβάνω, στηρίζουμε την πρόταση παρόλο που κάποια σημεία μας διεξαρεστούν, παρόλα αυτά νομίζω ότι ο τελικός απολογισμός είναι ότι γίνονται κάποια βήματα προς το εμπρός. Εσύ, Κύριε Άνστ, δέχεστε να σας υποβάλει μια ερώτηση, κυρία Σλέτ. Ναι, μπορείτε να υποβάλλετε την ερώτηση. Εντάχει, όπως ορίζει ο κανονισμός. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα γιατί η πολιτική σας ομάδα δεν κατέθεσε τροπολογίες στην Ολομέλεια που είχατε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό. Θα μπορούσατε να είχατε πετύχει τελικά το 100% χρηματοδότηση από το Συμβούλιο. Γιατί δεν το κάνατε. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν θεωρήσαμε ότι θα είχαν ελπίδα αυτές οι τροπολογίες, γι' αυτό και δεν τις καταθέσαμε. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν μας είχε αρέσει ιδιαίτερα. Όμως, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων έμαθα πολλά και διαπίστωσα διαπίστωσα ότι τελικά δεν ήταν τόσο καλή η πρόταση όσο θεωρούσαμε αρχικά. Επαναλαμβάνω, ναι θα μπορούσαμε να είχαμε καταθέσει τροπολογίες αλλά θεωρήσαμε ότι δεν θα είχαν καμία ελπίδα. Ο κύριος Βανίστερο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε εξαιρετικούς καιρούς χρειάζονται εξαιρετικά μέσα. Πρόκειται για κάτι που ζητούμε εδώ και πολύ καιρό, την απλούστευση ενός συστήματος για να αποδίδει περισσότερο και εντάχει. Αυτή τη βδομάδα έχουμε δημοσίευση αριθμητικών στοιχείων για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η πολιτική συνοχής. Μιλάμε για δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, μια πιο απλουστευμένη πολιτική όχι μόνο υπέρ των μεγάλων προγραμμάτων αλλά και των μικρών για τις ΜΜΕ, νέες τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Το θέμα της συγχρηματοδότησης δεν μας βρήκε σύμφωνους. Θα πρέπει να μην υπάρχει αυτός ο συγκεντρωτισμός και όλα τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν έτσι ώστε να προωθήσουμε περισσότερο την περιφερειακή ανάπτυξη. Και ένα άλλο σημείο είναι το εξής. Για μία πιο παρατεταμένη περίοδο να υπάρχει συγχρηματοδότηση και αν υπάρχουν καθυστερήσεις να πρέπει να προωθήσουμε αυτά τα σχέδια έτσι ώστε να μην χαθούν τα κονδύλια. Το... Από το 2007 το κάνουμε αυτό και ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο κατά πόσο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το καλό παράδειγμα και το 2008, 2009 και 2010. Ως προς το θέμα της αλληλεγγύης υπάρχουν ε, χώρες που δεν χρησιμοποιούν τα περιφερειακά ταμεία. Δηλαδή έχουμε 30 με 40% μη απορροφημένα κονδύλια. Τι θα γίνει με αυτά. Δεν μπορούμε να ορίσουμε έναν κοινό κορπανά σε αυτή την περίπτωση. Βεβαίως τρέχει ο χρόνος, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα εξορροπημένο σύστημα μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να φτάσουμε σε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο δώσω το λόγο στην κυρία Περβάνς Περές, την οποία δεν βλέπω όμως. Όμως βλέπω τον κύριο Γκάλαχερ, ο οποίος έχει και το λόγο για δύο λεπτά. Από το 73 και τούδε Έχουμε λάβει 80 εκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία. Με το πέρασμα του χρόνου αυτό διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Ιρλανδίας. Και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ιδιαίτερα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ιρλανδία για να καταπολεμήσουμε την ανεργία στην Ιρλανδία και στην Ευρώπη γενικότερα. Από το 1973 7 δις έχουμε λάβει από το κοινωνικό ταμείο, από το ΕΚΤ, για να αντιμετωπίσουμε τη μακροχρόνια ανεργία. Και υπό το πρόγραμμα ανθρωπίνων πόρων για την περίοδο 2007-2013, το Ευρωπαϊκό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας δώσει 377 εκατομμύρια δυνάμει του ΕΚΤ. Μιλάμε για 1,36 δις συνολικά για κατάρτιση των μη απασχολούμενων, για ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες και για ε, αυτούς που ε, έχουν που πρέπει να ανταποκριθούν σε ειδικέ περιστάσεις. Μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δράση του ΕΚΤ που βοηθά στην κατάρτιση, στη διαβίου κατάρτιση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Στα πλαίσια αυτή της χρηματοπιστωτικής κρίσης βλέπουμε ότι θα χρειαστούμε την υποστήριξη αυτού αμείου, ιδιαίτερα του ΕΚΤ. Ευχαριστούμε τους συνάδελφους. Η ε, κυρία Σουίμπερ, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση βασικά θέτει ορισμένους κέριους στόχους. Τα κράτη-μέλη που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τη χρηματοπιστωτική κρίση πρέπει να βρουν έναν τρόπο αντιμετώπισης. Και όλοι ζητούν κάποια βοήθεια για την εξισορρόπηση των προϋπολογισμών τους. Είναι σωστό μέτρο η προχρηματοδότηση των οικονομιών αυτών που προτείνεται. Τα κράτη-μέλη, πολλά κράτη-μέλη έχουν έλλειμμα 10% και παραπάνω. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει, αλλά η έκθεση αυτή δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Η ιδέα ότι τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να συγχρηματοδοτούν προγράμματα με από δικά τους χρήματα είναι πολύ επικίνδυνη ιδέα μπορεί να είναι σωστή για να εξισορροπήσει αλλά μας απαγορεύει να αναλάβουμε σημαντικά πράγματα. Δεν πρέπει λοιπόν να γίνει κατάχρηση της ιδέας αυτής, πρέπει απλώς να απλοποιηθούν οι κανόνες της χρηματοδότησης. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια την Ουαλία δεν πρόκειται να έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν έχει καμία τοπική αρχή χρήματα για να δώσει για χρηματοδότηση. Σωστό μπορεί να είναι να διαπιστώνουμε ότι οι πτωχότερες χώρες μέλη πρέπει να βοηθηθούν. Παρόλα αυτά και σε πλουσιότερες χώρες υπάρχουν περιφέρειες όπως η δική μου η που μπορούν να συγκριθούν με την οικονομική κατάσταση της Ρουάνδης. Μπορεί λοιπόν τέτοιου είδου ιδέες να καταλήξουν στην περαιτέρω υποβάθμιση περιφερειών σαν την Ουαλία και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Ευχαριστούμε κύριε Σουίνμπουρν. Για δύο λεπτά ο κύριος Κοβατσέφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κυρίλοφ για την έκθεσή του όταν έρθει θα τον συγχαρώ γιατί υποστηρίζω όλες του τις προτάσεις για τη διευκόλυνση της χρήσης των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων των Ελληνικής. Δεν μπορεί η Ένωση να εξομοιωθεί στα μάτια των πολιτών με, με το ηφαίστειο που γνωρίζετε που σκορπάει παντού στάχτη στα μάτια των πολιτών και τους αποκλείει από την πραγματοποίηση των προσδοκιών τους γιατί υπάρχει μια πραγματική δυσκολία στην απορρόφηση των διαρθρωτικών ταμείων. Γι' αυτό η απλοποίηση των διαδικασιών δεν είναι καθεαυτή κάτι το θετικό. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα και τον στόχο η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο με τις προτάσεις τους θα επιτρέψουν τελικά την ωφέλεια από τους τελικούς χρήστες. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των τροπολογιών, ορισμένων τροπολογιών, ιδίω μίας που θα επέτρεπε μακρύτερη περίοδο για τη δαπάνηση κονδυλίων που ενεκρίθησαν από το 2007 για να μπορέσουν χώρες με χαμηλό βαθμό απορροφητικότητας όπως η Βουλγαρία να δαπανίσουν χρήματα που αλλιώς θα χάνονταν και πρέπει όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες, μέλη, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που τους δίνεται με αυτή την τροπολογία. Η έκθεση τελικά νομίζω βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση γενικότερα ως προς την πολιτική συνοχή, αλλά συγκεκριμένα για την απλοποίηση των κανόνων. Επίσης πρόκειται για ένα βήμα προς τα εμπρός γιατί η έκθεση επιζητά μεγαλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ συντονισμού και ελέγχου. Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι εργαλείο για περισσότερη διαφάνεια για τον Ευρωπαίο πολίτη και φορολογούμενο καθώς και φορολογούμενη. Και πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν καθήκοντα που να είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν ώστε να μην καταστραφεί η οικονομική συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Ταμπατζή. Ευχαριστώ. Από, από τότε που ξέσπασε η κρίση ακούστηκαν επικρίσεις για, κατά της Ένωσης ότι λέει απέτυχε να, την αντιμετωπίσει. Η έκθεση αυτή όμως δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματι σε θέση να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους κρίσεις. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί ορισμένοι συνάδελφοι να λένε ότι η απλοποίηση μπορεί να καταλήξει σε κατάχρηση. Δεν συμφωνώ. Η πολιτική συνοχής είναι κάτι που υπονοεί και έναν αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, προϋποθέτει. Επομένως δεν θέλω να επιδεικνύουν αυτή την έλλειψη αλληλεγγύης ιδιαίτερα ως προς την Ουγγαρία. Η σωστή χρήση αυτών των κανόνων δεν δημιουργεί καμία κατάχρηση. Χρειάζεται η πολιτική συνοχή είναι χρήσιμη και θα ήθελα να πω στους ε, παρόντες επιτρόπους εδώ ότι ο κύριος Μπαρόσο μας είπε λίγα στις προγραμματικές δηλώσεις της Κομισιόν για την πολιτική συνοχή και παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικά κοινοτικά προγράμματα και μάλιστα θα έλεγα απαραίτητα για να μπορέσουν να δημιουργηθούν, να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης και να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι της Ένωσης, οι στόχοι του 2020. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Με όλες τις αλλαγές που έχουν ε, επέλθει στο διαρθρωτικό αυτό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας, δεν πρέπει να μας ε, κάνουν να ξεχνάμε ότι η υψηλή ανεργία έχει ε, ζωφρές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Αυτό που έχει σημασία είναι να εφαρμόσουμε πραγματικές πολιτικές σε συνοχή σε όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πραγματική ε, οικονομία μέσα με 347 δις ευρώ. Για αυτή την περίοδο θα πρέπει να, δοθεί περισσότερη, να δοθούν περισσότερα κονδύλια μέσα στα πλαίσια χρηματοδοτήσεων των περιφερειών των κρατών μελών. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια των, των επιμέρους ε, projects. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν και ήταν ένα ε, πολύ αναμενόμενο, ε, μια πολύ αναμενόμενη έκθεση, ε, δυστυχώς αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις όπου πολύ καλά μέτρα καθυστερούν. Θα πρέπει να πλουστεύσουμε το γραφειοκρατικό φόρτο για να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης και σε χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, όπως τη δική μου, τη Ρουμανία. Όπως ξέρετε, σε πέντε μέρες ανατράπηκαν τα πράγματα εξαιτίας της έκρηξης ενός ηφαιστείου πώς θα μπορέσουμε και πότε θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις με μεγαλύτερη σπουδή από εδώ και στο εξής. Ευχαριστώ. Η κυρία Σμόλκοβα, για να μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Λόβα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 ένα πρόβλημα με τη γλώσσα σας. Μπορείτε να επαναλάβετε. Μπορείτε να επαναλάβετε. Δεν ακούγαμε την διερμηνία στα αγγλικά. Έχει λυθεί όμως τώρα το πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ την εργασία του κ. Κυρίλοφ. Θα πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε σε μια τέτοια οικονομική κρίση και γι' αυτό απλουστεύουμε τη διαδικασία χρηματοδότησης περιφερειακών προγραμμάτων και απλουστεύουμε και τους κανόνες που διέπουν τα διαφορετικά ταμεία. Επίσης, οι προθεσμίες θα πρέπει να παρεκταθούν όπως ε, εγκρίθηκε το 2007 έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερη δυνατότητα χρήση στη Σλοβακία. Λέμε ότι όποιος χορηγεί γρήγορα είναι σαν να χορηγεί δύο φορές. Θα πρέπει λοιπόν έτσι να αντιμετωπίσουμε και τον υποεξέταση κανονισμό. Τον Ιούλιο πέρσι εισήχθη αυτός ο κανονισμός και η απόφαση θα ληφθεί το Μάιο. Χρειάστηκαν εννέα μήνες για αυτή τη διαδικασία. Ίσως θα πρέπει να απλουστεύσουμε την νομοθετική διαδικασία σε ορισμένες περιπτώσεις. Για την κρίση, ανεργία, φτώχεια, τις περιφερειακές ε, διαφορές θα πρέπει να δρούμε τάχιστα και με μεγαλύτερο δυναμισμό. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στους ανέργους ότι εμείς χρειαζόμαστε τρία τέταρτα του χρόνου για να εγκρίνουμε μια νομοθεσία, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση σε αυτό το γύρο ομιλητών. Η κυρία Γκρουνή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ομόφωνα σήμερα στηρίζουμε την απλοποίηση για τα διαθρώτικα ταμεία που προτείνει ο κύριος Κυριλόφ. Ωστόσο, ως υπεύθυνη για θέματα κοινωνικού ταμείου στο Κοινοβούλιο έχω κάποιες επιφυλάξεις. Καταρχάς να πω ότι είχαμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν τον Ιούνιο του 2009. Ο στόχος αρχικά ήταν η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκαν έξι μήνες για να κάνει κάτι το Συμβούλιο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σήμερα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτή την καθυστέρηση στους πολίτες μας. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δείξει υπευθυνότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έρθει πιο κοντά στη θέση του Συμβουλίου προκειμένου να μην καθυστερήσει περισσότερο η διαδικασία απόφασης με το Συμβούλιο. Πρέπει να λαμβάνουμε ταχύτατα αποφάσεις προκειμένου να έχουμε άμεσες επιπτώσεις επιτόπου. Η πρόταση σήμερα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έχει θετικά στοιχεία. Ωστόσο θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο φιλόδοξη, ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την περίοδο προγραμματισμού του 2007-2013, όπου τα πράγματα δεν ήταν τόσο δύσκολο. Για τον ε, νέο προγραμματισμό, για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2014-2020, θα ήθελα να ζητήσω μεγαλύτερη τόλμη από το Κοινοβούλιο προκειμένου να καταλήξουμε σε μεγαλύτερη απλοποίηση των διαδικασιών. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Έχουμε τέσσερις ε, υποψηφίους που προσέλκυσαν την προσοχή μου. Ο κύριος Σιλβέστρης είναι ο πρώτος και θα σας διακόψω στο λεπτό. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι ότι δέχομαι ε, το ότι ο κύριος Κυρίλοφ έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Λυπάμαι που δεν ήταν παρόν σήμερα. Θα πρέπει να ε, συνδράμουμε στο έργο του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διότι πρόκειται για διαρθρωτικά ταμεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όμως, θέλουμε ένα άλοθη για τις περιφέρειες, διότι δαπανούν αυτά τα χρήματα, αλλά δεν τα απορροφούν όλα, γιατί δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Αλλά μας... Ε, τι μας κάνουν, μας κατηγορούν ότι εμείς προβάλλουμε γραφειοκρατικά προσκόμματα. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και σας διακόπτω, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Ένσιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τα, ε, η κρίση, μάλλον η χρηματοοικονομική ε, κρίση, είναι απότοκη μιας κατάστασης άκρατης φτώχειας. Έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσουμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η έκθεση Κυρίλοφ η οποία, η οποία είναι ευπρόσδεκτη, διότι θα πρέπει να πλουστεύσουμε την διαδικασία πρόσβασης των κρατών μελών. Υποστηρίζω τα μέτρα που προτείνει ο κύριος Κυρίλοφ και από πλευράς προσαρμογής κριτηρίων για την βελτίωση της διαχείρισης. Αυτές οι τροποποιήσεις συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2010 που ενθαρρύνει την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ευχαριστούμε. Κυρία Τζεντεριεύσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπα, κυρίες και κύριοι. Οι προηγούμενοι μίλησαν για τα ωφέλη της πολιτικής συνοχής. Δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η περιφέρειά μου στην Πολωνία επίσης επωφελήθηκε από την πολιτική και από τα κονδύλια αυτά και χαίρομαι που βλέπω μια συνεχή προσπάθεια για μεγαλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει συνεχώς να απλοποιούμε τις διατάξεις και να τις κάνουμε πιο ευέλικτες. Πιστεύω λοιπόν ότι και ο κανονισμός αυτός θα αποτελέσει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και χαίρομαι γι' αυτό. Όμως επαναλαμβάνω ότι πρέπει να συνεχίζουμε συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική συνοχή είναι ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο που μας επιτρέπει να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης, στην αύξηση βραχυπρόθεσμα της ζήτησης και μακροπρόθεσμα στην αύξηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητάς μας. Η πολιτική συνοχής και η πληρωμές, η επιτάχυνση για το 2009 βοήθησαν πολύ προκειμένου να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη και να βελτιωθεί η ιδιωτική ζήτηση. Είναι λοιπόν σημαντική η συνεισφορά της πολιτικής συνοχής και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και το 2020. Να πω εδώ ότι ο Επίτροπος Όλη Ρεν στο θέμα των κυρώσεων για τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται τις κανόνες αγοράς θα ήθελα να έχει περισσότερες περιορισμούς στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που θα εγκριθεί άμεσα η έκθεση Κυριλόφ. Οι συμπολίτες μας ζητούν συγκεκριμένα μέτρα κατά της ε, κρίσης και οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες θέλουν περισσότερη ευελιξία στο θέμα της κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τώρα συζητάμε μέτρα για μεγαλύτερη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά κονδύλια συνοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η έκθεση Κυριλόφ είναι το πρώτο βήμα για μια απλοποίηση, αλλά χρειάζονται και άλλα. Γιατί η αξιοπιστία και η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή ζωή είναι κάτι πολύ σημαντικό που τίθεται ένα αμφιβόλο. Θα πρέπει να βρούμε μέτρα προσαρμογής στις νέες καταστάσεις. Θεωρώ ότι η έκθεση Κυριλόφ είναι μία ανάσα και ελπίζω όμως ότι δεν θα είναι παρά το πρώτο βήμα. Τελειώνουμε και με τις παρεμβάσεις αυτές και θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Χάν για να αντιδράσει στα λεγόμενα των ομιλητών κατά τη διάρκεια της συζήτησης ευχαριστώ κύριε πρόεδρε κυρίες και κύριοι. θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ενεργό ενδιαφέρον που δείξατε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί βλέπω σημαντική στήριξη, ευρεία στήριξη για την πολιτική συνοχή και βλέπω ότι διαπιστώνεται ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες των ασθενέστερων περιφερειών. Ο συνάδελφος από την Τσεχία μας είπε ότι όποιος δίνει γρήγορα προσφέρει τα διπλά. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σύνθημα για αυτόν τον κανονισμό Κυρία Σρέτερ, θα ήθελα να σας πω ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Δεν θα αλλάξουν οι έλεγχοι. Μπορεί να αυξήθηκε το όριο στα 50 εκατομμύρια για τα μεγάλα έργα, αλλά ακόμη και για τα μικρότερα έργα παραμένουν έλεγχοι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έχουμε εδώ να κάνουμε με την αρχή της ε, κοινής διαχείρισης. Και βεβαίως ε, παραμένει και η δέσμευσή μας για δημόσιους ε, διαγωνισμούς προκειμένου όλα να γίνονται με δημοσιότητα και διαφάνεια στο θέμα της ε, επιλογής έργων. Όσον αφορά τον κανονισμό και τον κανόνα νησιν 3, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περιοριστικοί εδώ ή και λιγότερο περιοριστική φτάνει να μην επιτρέψουμε στο σύστημα να κάνει κοιλιά. Θέλουμε οι περιφέρειες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια και να πω στην κυρία Σουίνμπερν ότι θεωρώ ότι έχουμε αρκετά κονδύλια για να συμπεριλάβουμε και την Ουαλία στην κατανομή κονδυλίων από το περιφερειακό και τα άλλα ταμεία. Και να πω ότι το σύστημα όσον αφορά την παραβίαση, τη μη συμμόρφωση συνήθως αποφεύγει τις οικονομικές κυρώσεις. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και ευχαριστώ και τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΡΕΤΖΙΟ της Επιτροπής. Η κυρία εξ ονόματος του εισηγητή. Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά θα διαβιβάσω τα όσα θετικά εκφράσατε προς τον κύριο Κύριλοφ. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα φορολόγησης. Θα πρέπει να είναι διαφανές το σύστημα, να έχουμε εύκολη, ε, καλύτερη προσπελασιμότητα. Και η κυρία Σρέτερ Κυρία Σέτερ, μη θεωρήσετε ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτά τα ευρωπαϊκά μέτρα. Είμαι πεπισμένος ότι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ε, αποδοτικά τα κονδύλια αυτά. Ε, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε και προς την κυρία Σουίνπερν βοηθάμε τις περιφέρειες έτσι ώστε να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία για να κινηθεί εκ νέου η ευρωπαϊκή οικονομία, ε, για να μπει σε τροχιά. Γνωρίζετε ότι είναι λογικό αυτό. Αυτή είναι μια σωστή οικονομική προσέγγιση, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα κονδύλια, για να χρησιμοποιηθούν ε, τάχιστα για να ανταποκριθούμε σε μια κατάσταση κρίσης. Ευχαριστούμε. Κλείνει και αυτή η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.